Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι γιατί μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που ε, θέμα έχει την προφορική ερώτηση για την θανατική ποινή. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην συντάκτρια της ερώτησης αυτής, την κυρία Ελένα Βαλενσιάνο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στις 10 του μηνός είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της ανητικής ποινής και είναι ε, επίκαιρο τώρα για να διατρανώσει η Ένωση τη διεθνή της δέσμευση υπέρ ενός παγκόσμιου μορατόριου των εκτελέσεων και να διατρανώσει τη θέση της για τη θανατική ποινή. Πού βρισκόμαστε. Υπάρχουν και καλά ναι λίγα μεν, αλλά πάρα πολύ άσχημα ναι Να αρχίσω από τα κακά νέα. Ακόμα 58 είναι οι χώρες που διατηρούν τη θανατική ποινή στην ένωμη τάξη τους. 22 από αυτές εκτελούν θανατικές ποινές, μάλιστα εκτέλεσαν το 2014. Ορισμένα κράτη επιβάλλουν τη θανατική ποινή σαν ισχυτικό αριθμό προσώπων είναι πολύ δύσκολο να φτάσουμε σε πληροφορίες και να τις συλλέξουμε γιατί υπάρχουν χώρες που δεν δίνουν στοιχεία για τις εκτελέσεις όπως είναι το Βιετνάμ και η Κίνα. Ε, ε, για παράδειγμα χώρες ε, πολύ σημαντικές και ουσιαστικά εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκρύπτουν στοιχεία που θα πρέπει εμείς κατηγορηματικά να ζητήσουμε γιατί επιπλέον η έλλειψη στοιχείων για την Κίνα ε, μας εμποδίζει να κάνουμε οποιαδήποτε στατιστική που να έχει κάποια αξία για να δούμε πώς επιβάλλεται η θανατική ποινή Αυτό είναι το πρώτο μου συμπέρασμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να απαιτήσει από τι χώρε με τι οποίε διατηρεί σημαντικέ σχέσει ακριβή στοιχεία για τον αριθμό των εκτελέσεων ε, σύμφωνα με ε, το πολιτικό και το στρατιωτικό τους νόμους. Οι εκτελέσεις ε, για τα μέρη του κόσμου όπου έχουμε στοιχεία μειώθηκαν με το 2014, 20% σε σχέση με το 2013 εκτελέσει, επαναλαμβάνω, για χώρε όπου έχουμε στοιχεία. Παρ' όλα αυτά, σε ορισμένε συγκεκριμένε χώρε οι εκτελέσει όχι απλώ δεν μειώθηκαν, αλλά αυξήθηκαν ε, το ίδιο διάστημα που μα απασχολεί. Το Ιράν έρχεται πρώτο με 229 εκτελέσεις που ανακοίνωσε το 2014 με δεύτερη την Σαουδική Αραβία ε, σε αυτό το Παλμαρές του Έσχους και ο πιο πολύτιμος μας ε, εταίρος, οι Ηνωμένε Πολιτείε 35 το 2014. Από τις 607 που εκτελέστηκαν το 2014, 70% ήταν σε τρεις μόνο χώρες. Ιράκ, Ιράν και Σαουδική Αραβία. Οι Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερικής, Ινδονησία, Ιαπωνία, Μαλαισία και Πακιστάν το 2014 εκτέλεσαν και ανθρώπους με αναπηρία σωματική ε, ή πνευματική. Το δεύτερο τμήμα της παρέμβασής μου θέλω να το αφιερώσω σε αυτό που αποκαλούμε το παγκόσμιο διάδρομο του θανάτου, δηλαδή εκείνους στους οποίους έχει επιβληθεί η θανατική ποινή αλλά δεν έχουν εκτελεστεί. Είναι οι Ε, 30% έχει αυξηθεί το 2014 η εκτέλεση. Άρα αυτός ο διάδρομος ανάτου παγκοσμίω δεν μειώνεται αλλά επιμικίνεται. Και επίσης πιστεύουμε ότι τα πραγματικά στοιχεία είναι πολύ υψηλότερα από αυτά που γνωρίζουμε. Η Αίγυπτος 509, Νιγηρία 659, Πακιστάν 231, και 142 στο Μπαγκλαντές. Αυτή είναι η πρώτη στις, ε, ε, στις καταδίκες το 2014. Αίγυπτος και Νιγηρία ε, έκρηξη σε αύξηση. Σας είπα, οι Ηνωμένε Πολιτείε επίσης 72 θανατικές καταδίκες το 2014. Παγκοσμίως πάνω από 19.000 ε, είχαν καταδικαστεί στη θανατική ποινή το 2014 και 8.500 ε, μόνο στο Πακιστάν ε, το οποίο ήρε το μορατόριο που είχε εξαγγελική και είχε δεσμευτεί η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και πολιτικές ομάδες ε, εντός αυτής κάνουν αυτή την προφορική ερώτηση. Σας ρωτάμε τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι μέτρα έχει λάβει για να προχωρήσουμε στην κατάργηση της θανατικής ποινής, ιδιαίτερα στις διμερείς σχέσεις με χώρες που τη διατηρούν και όπου αυξάνονται οι εκτελέσεις. Θα ήθελα να γνωρίζω επιπλέον μέχρι ποιου σημείου είμαστε διατεθειμένοι να φτάσουμε, μέχρι πού θα πιέσουμε ε, τα θεσμικά όργανα. Είμαστε διατεθειμένοι να θυσιάσουμε τις συμφωνίες που διαπραγματευόμαστε με κάποιες χώρες για να απαιτήσουμε μορατόριουμ και κατάργηση. Είμαστε διατεθειμένοι. Ε, είναι πολύ δύσκολο να συμφωνήσουμε με ορισμένες χώρες, αλλά ε, ορισμένες από τις χώρες είναι πολύ κοντά μας και έχουμε τις ίδιες αξίες και ιδέες, ας πούμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και νομίζω ότι νομιμοποιούμαστε να φέρουμε και ε, αυτό το θέμα πέρα από τις άλλες δυσκολίες που έχει η διαπραγμάτευση του TTIP. Δεν πρόκειται να σώσουμε ζωές εδώ. Δεν είναι μόνο αυτό. Να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να σωθούν αυτές οι ζωές και να ανταποκριθεί στη δέσμευσή της προς την κατεύθυνση αυτή και προς τις τρίτες χώρες. Επίσης, ευχαριστώ Πρόεδρο. Σας ευχαριστώ. Δέχεστε, κύριε Βαλασάνο, ε, μία μπλε κάρτα, ερώτηση με μπλε κάρτα από τον κύριο Κόρβιν Μίκε. Από ποιον? Από τον κύριο Κόρβιν Μίκε. Ε, Ας ε, συνεχίσουμε καλύτερα τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ για την ε, ξεκάθαρη και σταράτη απάντησή σας. Τώρα εκ μέρους του Συμβουλίου το λόγο έχει ο Υπουργό κ. Σμιτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη Ευρωβουλευτέ. Σας ευχαριστώ για την πολύ σημαντική αυτή ερώτηση που υποβάλλεται, γιατί η κατάργηση της θανατικής ποινής βρίσκεται στην καρδιά και είναι στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών αξιών. Κανένα κράτος δεν έχει το δικαίωμα να αποφασίζει ε, για τη ζωή, το θάνατο των πολιτών του. Όλοι πιστεύουμε ότι μία δίκαιη και απαραίτητη τιμωρία ποτέ δεν θα πρέπει να αποκλείει τη διάσταση ε, της ελπίδας και το στόχο της αποκατάστασης. Και αυτά είναι τα λόγια του Πάπα Φραγκίσκου στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά πρόσφατα. Από το 1983 το όχι στη θανατική ποινή αποτελεί τμήμα του κοινοτικού κεκτημένου είναι τμήμα της ταυτότητάς μας. Και αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που συμμετέχω σε αυτή τη συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λίγες μέρες πριν τη 10η Νοεμβρίου, την ε, Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής ποινής. Θα πρέπει να δώσουμε μάχη για να καταργηθεί η θανατική ποινή. Αξίζει αυτός ο αγώνας. Ας μην ξεχνούμε τη δική μας ιστορία. Ήδη, ήδη στη δεκαετία του 70 γινόταν ε, εκτελέσεις ακόμη και στη Δυτική Ευρώπη. Και θυμάμαι ότι σε μία από τις μεγάλες χώρες ένας σοσιαλιστής ε, πρόεδρος κατήργησε την θανατική ποινή το 1982. Πίσω από το σιδερό παραπέτασμα, μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 80 λάβανα χώρα θανατικές εκτελέσεις. Σήμερα όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απόλυτα απαλλαγμένη από τη θανατική ποινή. Βέβαια τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν και θα πρέπει εμείς να γίνουμε κινητήριος μοχλός της αλλαγής. Θα πρέπει να είμαστε όμως σαφείς και ξεκάθαροι ως προς ένα πράγμα. Και ποτέ να μην φοβόμαστε να διατρανώνουμε το στόχο της κατάργησης θανατικής ποινής ως τμήμα της εξωτερικής μας δράσης. Θα πρέπει να γίνει ακρογωνιαίος λήθος κάθε εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν από 10 χρόνια μόνο 59 χώρες είχαν πλήρως καταργήσει την θανατική ποινή. Τώρα έχουμε 101 χώρες. Πριν από 10 χρόνια, 41 χώρες ε, εκτελούσαν ακόμη θανατικές ποινές. Το 2014 μειώθηκε ο αριθμός στις 22, πολύ λιγότερες δηλαδή. Αλλά παρόλα αυτά και 22 είναι πολλές. Πολλές χώρες πρόσθεσαν τη θανατική τους ε, και την, και την εκτέλεσή της. Άλλες ε, μείωσαν την εμβέλεια των θανατικών ποινών. Σήμερα 140 χώρες ε, έχουν καταργήσει ε, de facto ή de jure τη θανατική ποινή. Βέβαια έχουμε και μια ζωφερή πλευρά στις στατιστικές πληροφορίες. Το 2015 είχαμε ακόμη χιλιάδες ανθρώπους που είτε καταδικάστηκαν σε θάνατο είτε εκτελέστηκαν. Ή χιλιάδες άνθρωποι είναι θανατοποινήτες παγκοσμίως. Ε, βέβαια, από το 2013 έχουμε είχαμε μείωση των θανατικών ε, ποινών, αλλά παρόλα αυτά ήταν, ε, είναι ακόμη τρομακτικά τα νούμερα, όπως ακούσαμε και από την κυρία Βελάνο. Η κατάργηση της θανατικής ποινής παγκοσμίω απαιτεί την κινητοποίησή μας, την ενέργεια και την πολιτική μας βούληση. Η χρήση της θανατικής ποινής για εγκλήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά είναι εμβληματική και αποτρόπαια πτυχή της χρήσης της θανατικής ποινής γιατί παγκόσμιο δίκαιο είναι σαφές. Τα εγκλήματα, τα συναφή με τα ναρκωτικά δεν είναι από τα σοβαρότερα εγκλήματα τα οποία θα μπορούσαν να επισύσουν και θανατική ποινή. Δυστυχώς πολλές ασιατικές χώρες εξακολουθούν να προβλέπουν θανατική ποινή για εγκλήματα ναρκωτικών. Στο Ιράν τουλάχιστον 75% από τις φετινές 660 εκτελέσεις ε, σχετίζονται με εγκλήματα για ναρκωτικά. Το ίδιο σχεδόν σε μικρότερη κλίμακα ισχύει και για τη Σαουδική Αραβία και για άλλες χώρες. Δυστυχώς όμως δεν είναι αυτό το μόνο ανησυχητικό στοιχείο και η μόνο ανησυχητική τάση. Εξακολουθεί να εφαρμόζεται θανατική ποινή για εγκλήματα που δεν ανήκουν στα σοβαρότερα κακουργήματα. Για παράδειγμα για οικονομικά εγκλήματα, για την αποστασία, τη ηχεία, ακόμη και τις σεξουαλικές σχέσεις ε, μεταξύ ενηλίκων που συνενούν. Και παρά τις ε, κατηγορηματικές ε, διεθνείς διατάξεις, μερικές χώρες εξακολουθούν να ανακαταδικάζουν και ακόμη και να εκτελούν ανήλικους ή πνευματικά καθυστερημένους. Δεν μπορούμε να αγνοούμε στην Ευρώπη το γεγονός ότι πολλές θανατικές ποινές είναι συνέπεια άδικων δικών χωρίς ε, εγγυήσεις ε, δικονομικές ε, και χωρίς τήρηση της αρχής της χάριτος. Επίσης χρησιμοποιούνται δημόσιοι αποκεφαλισμοί ή σταυρώσεις, αποτρόπες μέθοδοι δηλαδή, που επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τις οικογένειες των θανατοποιητών. Είναι αναφυσβήτο κύριε Πρόεδρε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ηγετικό ρόλο στην προσπάθεια κατάργησης της θανατικής πηγής. Η κατάργηση της θανατικής πηγής ε, εφαρμόζει σαφεί κατευθυντήρε γράμμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η μάχη μα κατά τη θανατική ποινή αποτελεί σημαντική προτεραιότητα και του νέου σχεδίου δράση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία που υιοθετήσαμε τον περασμένο Ιούλιο. Κατά το 2015 η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποίησε όλα τα διπλωματικά μέσα για να προωθήσει παγκοσμίω ε, την προσπάθεια κατάργησης της θανατικής ποινής. Και καταδικάζουμε ε, την εκτεταμένη χρήση της θανατικής ποινής ε, σε μερικές χώρες και μάλιστα ακόμη και γειτονικέ μας. Το Ιράν, το Ιράκ, η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν, η Ινδονησία, η Λευκορωσία, η Αίγυπτος, η Ιαπωνία, η Σιγκαπούρη, η Κίνα, το Βιετνάμ, Ακόμη και οι Ηνωμένε Πολιτείε, οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική ε, βρέθηκαν στο επίκεντρο της προσοχής μας. Πάνω από 30 δηλώσεις ε, ε, και διαβήματα έγιναν σε πολλές χώρες με βάση τις ελάχιστες προδιαγραφές που ορίζει το Διεθνές Δίκαιο και οι Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Γραμμές για τη θανατική ποινή. Ήμασταν οι πιο φανατικοί υπέρμαχοι της κατάργησης της θανατικής ποινής παγκοσμίω. Βέβαια, μερικοί από εσάς ε, ξεκολουθείτε να πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν τόσο, δεν τόσο σεντόρια τη φωνή της όπως θα έπρεπε. Θα είμαι ειλικρινής. Ε, μερικές φορές δεν αρκούν δηλώσεις ε, και το καλύτερο είναι να δεσμευτούμε και να συνεννοηθούμε ακόμη και με εκείνους που δεν εστερνίζονται τις αξίες μας. Αυτή είναι η πιο σημαντική συμβολή που μπορούμε να προσφέρουμε για την κατάργηση της θανατικής ποινής. Γι' αυτό και ενισχύουμε το διάλογο μας και τον εντατικοποιούμε με τις ε, χώρες που εφαρμόζουν θανατική ποινή και μάλιστα το κάνουμε σε όλα τα επίπεδα. Και ενισχύουμε τις προσπάθειες, ακόμη και σε, ιδιαίτερα σε χώρες που έχουμε έξαρση των εκτελέσεων ή επανεισαγωγή της θανατικής ποινής μετά από δεκαετίες μορατόριου. Και μάλιστα στις ε, μεμονωμένες στρατηγικές ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τις διάφορες χώρες έχουμε θέσει ως ύψιστη προτεραιότητα της, ε, την κατάργηση της θανατικής ποινής. Και μάλιστα ε, στο διάλογό μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουμε μονίμως το θέμα της θανατικής ποινής στην ε, ημερήσια διάταξη. Ακόμη και όταν συζητούμε με χώρες που έχουμε παρόμοιες ιδέες όπως είναι η Ιαπωνία, οι Ηνωμένε Πολιτείες. Το θέμα της θανατικής ποινής πάντως το θέτουμε όλες ε, τις διαπραγματεύσεις πέρα στρατηγικών συμφερόντων. Μιλούμε με το Πακιστάν, το Ιράν, τη Σαουδική Αραβία, αλλά και άλλες χώρες, ε, επισημένοντας ότι δεν είναι ε, φάρμακο, δεν είναι τιμωρία για τρομοκρατία, ναρκωτικά ή άλλα εγκλήματα συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας και τη δεσμευσή μας. Και οι διμερείς σχέσεις δεν είναι η μόνη ευκαιρία για να ευθέσουμε το θέμα αξιοποιούμε και τις περιφερειακές συναντήσεις. Για παράδειγμα, στην Αφρική έχουμε τη μεγαλύτερη συγκέντρωση χωρών όπου ε, υπάρχει μεγάλο δυναμικό ε, κατάργηση θανατικής ποινής για να γίνει και η Αφρικανική Ήπειρος η δεύτερη Ήπειρος που θα είναι απαλλαγμένη από θανατική ποινή. Γι' αυτό και στηρίζουμε τις πρόσφατες πρωτοβουλίες της Αφρικανικής Ένωσης για τη θέσπιση συμπληρωματικού πρωτοκόλου στο Αφρικανικό Χάρτη για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των λαών, προβλέπει η κατάργηση θανατική ποινή. Επίση, οργανώνουμε εκστρατείε στι ασιατικέ χώρε, προκειμένου να τροφοδοτήσουμε τη δημόσια συζήτηση για το θέμα του δικαιώματος στη ζωή και στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Επίσης, ε, συνεργόμαστε στενά με την ε, Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και ιδιαίτερα στο ψήφισμα για το μορατόριο των θανατικών εκτελέσεων. Και χάρη στις πιέσεις μας, ε, το μορατόριο υιοθετήθηκε το Δεκέμβριο του 2014 με 170 ψήφους υπέρ, άνευ υποστήριξη και 95 ε, ε, χώρες που μας υποστήριξαν στην προσπάθεια. Θέλουμε φυσικά εταιρικέ σχέσεις και σε παγκόσμιο επίπεδο για να επιτύχουμε στον αγώνα μας. Και η επιτυχία μας για το μορατόριο μας δίνει το μήνυμα ότι δεν είμαστε μόνοι στον αγώνα αυτό. Θα ήθελα κύριε Πρόεδρε να εκφράσω επ' ευκαιρία την ευγνωμοσύνη μου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την θερμή υποστήριξη ε, του αγώνα της καταρρής θανατικής ποινής. Αυτό φάνηκε σε αναρρύθμιτα ψηφίσματα σχετικά, αλλά και σε αποστολές σε τρίτες χώρες, όπου ευρωβουλευτές ε, δεν φοβούνται να θέσουν το ζήτημα των ε, εκτελέσεων, ακόμη και με τους πιο δύσκολους συνομιλητές μας. Επίσης έχουμε ένα παγκόσμιο δίκτυο εταίρων η πρόθεση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και το παγκόσμιο μορατόριο για τη θανατική ποινή βρίσκεται στην καρδιά και της εξωτερικής μας πολιτικής. Βρίσκεται στα θεμέλια και ανήκει στις θεμελιώδες αξίες και αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα συνεχίσουμε τις ε, συνομιλίες με τους εταίρους μας ε, ε, για το θέμα αυτό, για να έχουμε ένα πλανήτη στον οποίο καμία χώρα δεν θα είναι κυρίαρχος και δεν θα αποφασίζει για τη ζωή και το θάνατο των πολιτών της. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα να σας ενημερώσω αγαπητοί συνάδελφοι ότι η διαδικασία της μπλε κάρτας δεν ισχύει απέναντι στους εκπροσώπους του Συμβουλίου. Ισχύει μόνο μεταξύ των Ευρωβουλευτών. Τώρα θα δώσω το λόγο στους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων, αρχής γενομένης από τον κυρίο Αντάκτουσον, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ευχαριστώ πολύ. Η Διεθνής Αμνηστία μας λέει πως οι περισσότερες εκτελέσεις γίνονται στην Κίνα αυτή τη στιγμή. Και μετά ακολουθούν το Ιράν και η Σαουδική Αραβία. Στη Σαουδική Αραβία οι εκτελέσεις θεωρούνται ως ο μοναδικός τρόπος δημόσιας διασκέδασης μαζί με τους παιδοσφαιρικούς αγώνες και οι εκτελέσεις αυτές είναι σταυρώσεις, αποκεφαλισμοί, σύμφωνα με τον Ισλαμικό νόμο. Νομίζω ότι μιλάμε για μία εικόνα βαρβαρότητας, αλλά δεν μπορούμε να απλουστεύουμε τη συζήτηση για τη θανατική ποινή εξετάζοντας μόνο το πώς εκτελείται αυτή. Μιλάμε για ανθρώπινη αξιοπρέπεια και βασιζόμενη στις ε, χριστιανικές και ιουδαίκες ε, παραδόσεις στις οποίες βασίζονται οι δικές μας κοινωνίες θα πρέπει οι άνθρωποι να ζητούν άφεση για τα εγκλήματά τους και μετά να τους προσφέρεται ε, συγχώρεση γιατί το αδίκημα θα πρέπει να τιμωρείται όχι το άτομο και βέβαια η θανατική ποινή καταστρατηγεί αυτή την αρχή και κατά της αρχής του δικαιώματος στη ζωή στις 10 Οκτωβρίου είναι η 13η ημέρα δράσης κατά της θανατικής ποινής. Είναι μια ευκαιρία να τονίσουμε τις αξίες στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι αξίες αυτές θα πρέπει πάντα ε, να στηρίζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Εκ μέρους των σοσιαλιστών θα δώσω το λόγο στον κύριο Παντσέρη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η θανατική ποινή είναι η πιο απάνθρωπη τιμωρία. Το δικαίωμα στη ζωή είναι θεμελιώδες και μιλάμε για μια βίαιη τιμωρία η οποία δεν μπορεί να λαμβάνει χώρα ε, στο πλαίσιο της σημερινής απόδοσης δικαιοσύνης. Πολλές χώρες δικαιολογούνται λέγοντας πως αποτρέπει τα άτομα από το να εγκληματίσουν, πως είναι ε, δικαιώματα και κακοργήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά, πως στηρίζει η κοινή γνώμη, πως είναι θέμα εγκληματικότητας και πολλοί πιστεύουν πως το να καταργήσει κανείς τη θανατική ποινή θα αυξήσει τον αριθμό των ατόμων που εγκληματών. Το... Πρέπει να σας πω πως σε χώρες που κατάρρισαν τη θανατική την θανατική ποινή μειώθηκε και ο αριθμός των βίων ε, δολοφονιών. Μιλάμε για μία ε, ακραία ε, κύρωση που μπορεί να επιβάλλει ένα κράτος σε ένα άτομο χρησιμοποιώντας την βία και επαναλαμβάνοντας τον κύκλο της βίας αυτής. Οι εγκληματίες όταν ξέρουν ότι αντιμετωπίζουν τη θανατική ποινή δεν έχουν κανένα λόγο ε, που να τους αποτρέπει από το να ε, διαπράξουν και άλλες δολοφονίες. Για παράδειγμα, αν κάποιος επιτεθεί για να ληστεύσει μια τράπεζα και ξέρει ότι μπορεί να, κατα, ε, να καταδικαστεί στη θανατική ποινή, μπορεί να δολοφονήσει και δύο-τρεις από αυτούς που θα βρει στο διάβα του. Όταν έχουμε λοιπόν αδικήματα που συνδέονται με τα ε, ναρκωτικά, τα οποία καταδικάζουν σε θανατική ποινή, στη Μαλαισία, στη Σιγκαπούρη, στην Κίνα, στην Ινδονησία, χωρίς τα τεκμήρια και τα αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι αποτρέπουν με τον τρόπο αυτό ε, ε, από τους εγκληματίες, περισσότερο για παράδειγμα τους καταδίκαζαν σε μία ποινή κάθεξης πολιετή είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία θα πρέπει να πριτανεύσουν και θα πρέπει να εξηγήσουμε χώρε αυτές για ποιο λόγο αυτού του είδου η θανατική ποινή δεν δικαιολογείται. Η, η Διεθνής Αμνηστία ε, λέει πω η στήριξη από την κοινή γνώμη στη θανατική ποινή βασίζεται στην επιθυμία των ανθρώπων να μην υπάρχει έγκλημα στην κοινωνία. Αλλά έχουμε μελέτε που αποδεικνύουν πω. Όταν προτάθηκε η διαβίου κάθεξη για τέτοιου είδου εγκλήματα, η στήριξη για την εθνική ποινή σε κάποιε περιπτώσει μειώθηκε κατά 65%. Και ξέρετε πόσο κοστίζει να ε, θανατώσει κανείς κάποιον ε, ε, γιατί έχουν χρησιμοποιηθεί και οικονομικά και οικονομικές δικαιολογίες λέγοντας πως έχουν γεμίσει φυλακές και το κόστος διατήρησης κρατουμένων είναι τόσο υψηλό που θα πρέπει να προχωρήσουμε σε εκτελέσεις. Αυτά τα πράγματα είναι ανεπίτρεπτα. Δεν θα αλλάξουμε την κατάσταση στις φυλακές μέσω τη θανατικής ποινής. Α πούμε όχι στη θανατική ποινή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δράσει με αποφασιστικότητα έτσι ώστε να καταργηθεί παντού. Ευχαριστώ στη ο κύριος Μάρκ μέσμακερ για ένα λεπτό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, κάθε εκτέλεση με σκοτώνει. Κάθε εκτέλεση είναι μια ήττα και μια απόδειξη ανικανότητας. Ήττα για την ανθρωπότητα ολόκληρη και για την ανθρωπιά. Είναι η ανικανότητα να επιβάλλει το δίκαιο με έναν τρόπο ε, ανθρώπινο και όχι βάρβαρο ε, ανέντιμο. Είναι γεγονός ότι παγκοσμίω έχουν μειωθεί οι εκτελέσεις και πολλές ε, χώρες την κατήργησαν τη θανατική ποινή τα τελευταία χρόνια. Αλλά απέχουμε πόρο από παγκόσμια κατάργηση. Και σε κάποιες χώρες είναι αποτρόπαια τα στοιχεία. Πολλές φορές είναι και κρατικό μυστικό. Αλλά γνωρίζουμε για παράδειγμα ότι το Ιράν και μόνο στο πρώτο εξάμεινο του 2015 εκτέλεσε 600 ανθρώπους και συχνά για μη βία ε, εγκλήματα όπως για μοιχεία ή άλλα εγκλήματα σχετιζόμενα με ναρκωτικά. Και σε άλλες χώρες η κατάσταση είναι ανισχυτική. Και χαίρομαι για την πρωτοβουλία στα Ηνωμένα Έθνη της ε, Ομοσπονδιακής μου κυβέρνησης να επανέλθει το θέμα στη διεθνή ατζέντα. Αν ε, το Συμβούλιο ε, θέλει να δώσει μεγαλύτερη σημασία στο θέμα, το ενδιαφέρουν όχι μόνο τα οικονομικά αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τότε θα βρει στο Κοινοβούλιο πλήρη υποστήριξη προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα εξ ονόματος των φιλελευθέρων το λόγο έχει η κυρία Μπεατρίθ Βεθέρα Μπαστερετσέα. Για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η θανατική ποινή είναι ίδιον ε, της βαρβαρότητας, έλεγε ο Βίκτορ Ουγκό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ε, ορίζεται από τις αρχές και δημοκρατικές αξίες. Θα πρέπει να είμαστε πρωταγωνιστής για να τερματιστεί η θανατική ποινή σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορούμε να ανεχθούμε τη βαρβαρότητα. Και τώρα που γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα θα πρέπει να ε, δώσουμε ένα παράδειγμα σε εκείνους που το 2014 καταδίκασαν σε θάνατο 2.500 ανθρώπους και θα πρέπει να είμαστε υποδειγματικοί και για τους ίδιους. Πουθενά δεν θα πρέπει ε, σε καμία περίπτωση στην Ευρώπη να εξετάζει κανένα κράτος το ενδεχόμενο να επαναφέρει τη θανατική ποινή. Αυτό θα παραβίαζε τις συνθήκες και το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Το εγχείρημα αυτό είναι πολύ βασικό και δεν μπορούμε μόνοι μας να το κάνουμε. Χρειαζόμαστε στο πλευρό μας τις Ηνωμένε Πολιτείε για να τερματιστεί εκεί. Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, Κίνα, Ιράν και Σαουδική Αραβία πρωτοστατούν ε, στις εκτελέξεις. Στην ε, Κίνα παραμένουν κρατικό μυστικό οι ε, αριθμοί. Σαουδική Αραβία εκτελούν δημόσια. Ο Αλή Αλ Νίμρ, 17 ετών, το συνέλαβαν γιατί αγωνιζόταν για την δημοκρατία και έχει καταδικαστεί ε, να ε, τον αποκεφαλίσουν. Ε, για, να σας μιλήσω για το Ιράν. Η λεγόμενη μετριοπαθής κυβέρνηση του Ρουχανή εκτελεί τρεις ανθρώπου τη μέρα, γύρω στους 700 το πρώτο εξάμεινο. Αν ρωτήσουμε την Αθηνά Νταεμή ή την Αθηνά Φαρχαδάνη δεν θα μπορέσουν να μας απαντήσουν. Είναι νέες Ιρανές που τις φυλάκισαν για κάποια σκίτσα στο διαδίκτυο ή κατήγγυλαν ε, τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από πλευρά κυβέρνηση Ιράν. Αν τις ρωτούσαμε όμως θα μας έλεγαν αν μπορούσαν ε, ότι αξίζει τον κόπο. Δεν μπορούμε να ανεχθούμε τη βαρβαρότητα σε καμία έκφανσή τη. Ε, και πιο είναι η θανατική ποινή. Δεν επιτρέπεται να τις απογοητεύσουμε αυτές τι κοπέλε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εξ ονόματο ε, της Κουατζέλ, η κυρία Βεριά. Για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχει καμία δράση που να είναι πιο βαρβαρική από, πιο βάρβαρη, με από τη θανατική ποινή. Είναι ένας παγκόσμιος αγώνας ο οποίος ακόμα δεν έχει ε, φτάσει στο τέλος του. Αυξάνεται ο ρυθμός των χωρών που την επιβάλλουν και η ΕΠΑ ε, είναι μια σκιά στις δημοκρατικές χώρες, μια και εκτελεί αυτές τις αποφάσεις. Έχουμε χώρες οι οποίες είχαν αποφάσει σε ένα μορατόριμο, όπως η Πακιστάν και η έχουν ξαναξεκινήσει. Η κατάργηση της θανατικής ποινής ε, έχει περιοριστεί και κάποιοι την έχουν επανεισάγει. Και μάλιστα πρέπει να σας πω πως αυξάνεται και ο ρυθμός εκτελέσεων και όχι μόνο στη Δική και στο Ιράν. Είναι η μάχη κατά της τρομοκρατίας και των ναρκωτικών που είναι το φιλουσικής που καλύπτει την επιβολή αυτών των θανατικών ποινών σε χώρες όπως η Αίγυπτος. Και πρέπει να σας πω ότι είναι αρκετές οι χώρες η Τουνησία για την οποία από το 1991 υπήρχε μορατόριο που ξανασκέφτονται το θέμα αυτό. Και πρέπει να σας πω πως οι δηλώσεις του κυρίου Όρμπαν το Μάιο είναι υπερβολικά πολλοί αυτοί οι οποίοι ε, προσπαθούν να ξανασυζητήσουμε το θέμα επειδή ε, ε, διακατέχονται από ένα κακό εννοούμενο λαϊκισμό. Δεν θα πρέπει ποτέ εμείς με τα δικά μας προγράμματα να χρηματοδοτούμε άμεσα ή έμεσα αυτές τις βάρβαρες πρακτικές. Θα πρέπει να σταθούμε άγρυπνα για να αποφύγουμε να συμβεί κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος τώρα των Πρασίνων, το λόγο έχει η κυρία Μπάρμπαρα Λόχπιλερ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η θανατική ποινή δεν είναι ανάλογη ε, στην εγκληματικότητα. Δεν μπορεί το κράτος να επιβάλλει το θάνατο. Αυτό δεν είναι δικαιοσύνη, είναι αντίπεινα και εκδίκηση. Αυτό φρονεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει ε, δεσμευτεί να αγωνιστεί για την κατάργηση ε, και με επιτυχία. 101 είναι οι χώρες που έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή για όλα τα κακουργήματα. 33 στην πράξη αλλά όχι στην νομοθεσία. Δυστυχώς σε κάποιες χώρες βλέπουμε δραστική αύξηση των εκτελέσεων και δυστυχώς 7 χώρες το 2014 άρχισαν να ξαναεκτελούν ε, μετά από μορατόριο ετών η θανατική ποινή σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο ε, μπορεί να επιβληθεί σε πάρα πολύ δεχθεί εγκλήματα. Σε 33 χώρες όμως εφαρμόζεται για ε, εγκλήματα που συνδέονται με τα ναρκωτικά όπως στην Κίνα, στο Ιράν και στη Σαουδική Αραβία. Και εδώ αγωνίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για να καταργηθεί η θανατική ποινή. Ταυτόχρονα όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη συμμετέχουν ε, με χρηματοδότηση στην καταπολέμηση των ναρκωτικών ε, μέσω των αντίστοιχων οργανισμών του ΟΗΕ. Η ανεξάρτητη έλεγχη στο Πακιστάν και το ε, Ιράν των προγραμμάτων αυτών αφήνουν να εννοηθεί ότι υπάρχει σχέση με την εφαρμογή της αντικής ποινή. Αυτό είναι ανησυχητικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να φροντίσει ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι προδιαγραφέ του να εφαρμόζονται παντού όπου υποστηρίζουμε προγράμματα κατά των ναρκωτικών και να έχουμε ενημέρωση. Γιατί η κατάργηση τη θανατική ποινή για ε, αδικήματα που συνδέονται με ναρκωτικά θα πρέπει να είναι προπόθεση και προαπαιτούμενο για τη χρηματοδότηση τέτοιων προγραμμάτων. Ευχαριστώ. Do Δέχεστε μια μπλε κάρτα από τον κύριο Κόρβιν Μίκε. Θα προτιμούσα να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Εκ μέρους της ομάδας EFDD, ο κύριος Άρνοτ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Δεν είμαι απαδός της θανατικής ποινής, αλλά είμαι απαδός της δημοκρατίας. Ακούσαμε την ε, τι απόψει κατά τη θανατική ποινή και μάλιστα επανειλημμένε. Και γενικώ συμφωνώ. Αν όμω ρωτούσα του ψηφοφόρου μου στην εκλογική μου περιφέρεια τη γνώμη του. μάλλον θα ήταν διχασμένε οι απόψεις. Ε, για, παράδειγμα, κάποιο ε, που βάναυσα ε, στερεί από κάποια τη ζωή, μήπω έπρεπε και αυτό να χάσει τη ζωή του. Επίσης, ε, το άδικο σύστημα της Σαουδαραβίας ε, δεν θα πρέπει να το καταδικάσουμε. Βέβαια. Όχι όμως για τη θανατική ποινή. Αλλά το θέμα αυτό είναι απόφαση μιας ε, κυρίαρχης κυβέρνησης. Το θέμα είναι ότι συστηματικά άδικα εφαρμόζεται το σύστημα. Φυσικά είμαι κατά της θανατικής ποινής, αλλά είναι λάθος να πολιτικοποιούμε μια συζήτηση επιβάλλοντας μια θέση έναντι άλλης και προβάλλοντάς την ως τη μοναδική έγκυρη θέση. Ευχαριστώ. Δέχεστε μπλε κάρτα από τον συνάδελφό σας, τον κύριο Παρακαλώ. Συνήθως ε, συμφωνούμε με τον κύριο Άρνοτ. Εδώ διαφωνούμε όμως. Συμφωνείτε κύριε Άρνοτ ότι, ε, ότι μερικά εγκλήματα μόνο ο Θεός μπορεί να τα συγχωρέσει. Ή συμφωνείτε ότι η συμφωνείτε ότι η πρωτοκαθεδρία της δημοκρατίας είναι ο σημαντικότερος παράγοντας σε κάθε έθνος κράτος και για κάθε πολιτικό. Αλλά αν ο λαός μιας χώρας με δημοψήφισμα δημοκρατικά ζητούν επαναφορά της θανατικής ποινής, νομίζω ότι κάθε πραγματικός και γνήσιος δημοκράτης οφείλει να δεχτεί αυτή την ετοιμιγορία. Εγώ πιστεύω στην αρχή της δημοκρατίας. Και ναι, αν ο λαός μιας χώρας θέλει να επαναφέρει τη θανατική ποινή, φυσικά θα πρέπει να το δεχτώ. Αλλά θα περίμενα και από τον κύριο Αθαρίς να δεχτεί ότι αν επικρατήσει ε, η δική μου θέση να δεχτεί να μην υπάρχει, να μην εφαρμόζεται θερατική ποινή. Αυτό είναι δημοκρατία. Αυτό θα πει δημοκρατία. Ε, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να δίνουμε την εξουσία σε ένα κράτο ε, για να αποφασίζει για τη ζωή το θάνατο των πολιτών. Δεν μπορούμε να ε, εικάζουμε ότι ένα κράτο έχει πάντα δίκιο. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Κομοντίνη Κάκια Τερέζα. Για 1,5 λεπτό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κατάργηση Θανατική ποινή είναι ουσιαστική για την προστασία τη ανθρώπινη αξιοπρέπεια και για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ας είμαστε σαφείς, όταν μιλάμε για κατάργηση της θανατικής ε, ποινής δεν λέμε πως θα μένουν ατιμόρυτα τα εγκλήματα. Χωρίς να μπαίνουμε στη συζήτηση με το κατά πόσο είναι ανάλογα με το έγκλημα τα, ε, οι, οι ποινές, υπάρχει ένα πιο ουσιαστικό θέμα που προκύπτει για την θανατική ποινή. Δεν μπορούμε να δεχτούμε την επιβολή μιας ποινής η οποία αποτελεί η ίδια καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Γιατί βέβαια καταστρατηγεί την ανθρώπινη αξιοπρέπεια στον ίδιο της τον πυρήνα και Βλέπει κανεί πως πολύ συχνά η θανατική ποινή ε, συνοδεύεται από συστήματα δικαιοσύνης που δεν μας εμπνέουν εμπιστοσύνη. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει εμείς να έχουμε μεγαλύτερη δέσμευση ε, υπέρ της κατάρρισης αυτής της ποινή. Είναι καλό που τα θεσμικά όργανα προσπαθούν να μας ευιστοποιήσουν για το θέμα αυτό με την ημέρα την οποία έχουν αφιερώσει στο θέμα. Αλλά χρειαζόμαστε πιο στεναρή δέσμευση και θα πρέπει η πολιτική μας συζήτηση να ενισχύσει την ε, ε, συζήτηση που γίνεται και να στηρίξουμε την κοινή γνώμη, να την ενημερώσουμε έτσι ώστε να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για να έχουμε και δικές δίκες αλλά και να καταργηθεί πατού η θανατική ποινή. thank you. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη, δέχεστε μια μπλε κάρτα από τον κύριο Κόρβιν Μίκε. No, Όχι, Πρόεδρε. Θα προτιμούσα να συνεχιστεί η συζήτηση. Ευχαριστώ. Ε, um, σας ευχαριστώ. Well, uh... Λοιπόν, και τώρα το λόγο. Ε, deputat Andy Christea. Κύριε αντι Christea. Για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για τα ρωμανικά σας κύριε Πρόεδρε. Η κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλα τα κράτη του κόσμου είναι από τους βασικούς στόχους της ε, πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τα πολιτικά και τα ανθρώπινα μάλλον δικαιώματα. Η θανατική ποινή βεβαίως είναι ασυμβίβαστη με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και σύμφωνα με έρευνες η θανατική ποινή δεν αποθαρρύνει τα βία εγκλήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος δωρητής στις προσπάθειες που κάνει η παγκοσμίωση κοινωνία των πολιτών και η παγκόσμια κοινότητα για να καταργήσει τη θανατική ποινή. Οι πρώτοι ήμασταν εμείς εκείνοι που ε, εισαγάγαμε κανόνες για να απαγορεύεται το εμπόριο στα διάφορα είδη συσκευέ ε, και προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση θανατικής ποινής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χρέος να ενθαρρύνει τον επικοδομητικό διάλογο για τα θέματα αυτά και να ε, ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη με εκστρατείες συνειδητοποίησης και ενημέρωσης. Θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να πείσουμε τις χώρες που εφαρμόζουν ε, θανατική ποινή να την καταργήσουν ή να προχωρήσουν σε δικαιοστάσιο. Ε, Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Βίξτρο. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τίποτα δεν είναι τόσο οριστικό ο θάνατος. Τίποτα δεν είναι τόσο μόνιμο και αμετάκλητο ο θάνατος. Και έχουμε σε πολλές χώρες απελευθέρωση φυλακισμένων μετά από πολλά χρόνια όταν έχει αποδειχθεί ότι φυλακίστηκαν ενώ ήταν αθώοι. Εδώ υπάρχει δυνατότητα επανόρθωση. Αν κάποιο όμω έχει καταδικαστεί σε θάνατο, σε περίπτωση που υπάρχει δικαστική πλάνη, δεν μπορεί να διορθωθεί αυτή η κατάσταση. Θα πρέπει να δώσουμε μάχη για να καταργηθεί η θανατική ποινή, που είναι, ε, δείχνει έλλειψη πολιτισμού, βαναυσότητα και από αποτρόπαια και ομή συμπεριφορά εκ μέρου του κράτου. Θα πρέπει αυτή να γίνει η προτεραιότητά μας. Θα πρέπει να συμβάλλουμε οπωσδήποτε στην κατάργηση της αναδυτική ποινή όπου και να εφαρμόζεται στον κόσμο. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριο Ευχαριστώ πολύ. Ξέρετε κι εσείς πως αύριο ο Ισπανός Βασιλιάς θα λάβει το λόγο εδώ στην Ολομέλεια και η δική του οικογένεια ε, έχει πολύ στενούς δεσμούς φιλίας με την βασιλική οικογένεια της Σαουδικής παραβίας, πρωταθλήτριας θανατικές ποινές. Μήπως δεν θα είναι άσχημο αύριο να του μεταφέρουμε την ανησυχία μας για τη θανατική ποινή και να του ζητήσουμε να επηρεάσει την Σαουδική Μοναρχία έτσι ώστε να τελειώσει και εκεί το θέμα της θανατικής ποινή. Είναι δύσκολο να με ακούσουν οι άλλοι οι Ισπανοί ε, βουλευτές εδώ γιατί δεν είναι στην αίθουσα, μάλλον δεν τους ενδιαφέρει η συζήτηση, αλλά νομίζω είμαστε όλοι κατά της θανατική ποινή. Άρα λοιπόν επειδή έχουμε πάρα πολλούς, υπερβολικά πολλούς εμπορικούς ε, εταίρους οι οποίοι εφαρμόζουν θανατική ποινή και επειδή είναι στον ΠΟΕ και τους υποχρεώνουμε να είναι στον ΠΟΕ, γιατί δεν τους υποχρεώνουμε να καταργήσουν και θανατική ποινή. Είμαστε οικονομικός γίγαντας. Γιατί να μην κάνουμε λιγότερες γιορτές και λιγότερες επαιτίους και να μην απαιτούμε από τους εμπορικούς μας εταίρους να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό ο κύριος Λαμπέρ. Κυρία, Κυρία Λαμπέρ. Όπως και εγώ καλωσορίζω τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της αναδικής ποινής, αλλά χρειαζόμαστε να έχουμε μια συνεκτική στάση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στις παρεμβάσεις που κάνει για τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορεί να είναι αποτελεσματική. Και κυρίως όταν έχουν γίνει στα πλαίσια διαπραγματεύσεων, οι οποίες για τις χώρες με τις οποίες διαπραγματευόμαστε έχουν σημασία. Για παράδειγμα, το γενικευμένο σύστημα προτιμήσεων ε, συν, ε, η ποιότητα της δικαιοσύνης που ανώμα, απονέμεται σε χώρες οι οποίες έχουν ακόμα τη θανατική ποινή πολλές φορές δεν είναι υπρέπουσα και η χρήση θανατικής ποινής σε κάποιες από τις χώρες αυτές είναι και πολιτικό εργαλείο. Όπως και άλλοι, λυπάμαι που το Πακιστάν έχει καταργήσει το δικαιοστάσιο στην ε, θανατική ποινή και έχει ξαναξεκινήσει τις εκτελέσεις και για κάποιους οι οποίοι δικάστηκαν υπό το καθεστώς Μουσαράφ και χαιρετίζω την αναστολή ε, για τον, Μπαζίτ, ε, στον, για τον κύριο Μπαζίτ στο Πακιστάν που αντιμετωπίζει σοβαρή αναπηρία και ελπίζω πως θα συνεχίσουμε στα πλαίσια του GSP Plus να ε, παρακολουθούμε τι γίνεται με αυτή την υπόθεση. Σας ευχαριστώ. Κοράω παρακαλώ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Είναι σαφές ότι η θανατική ποινή είναι η πιο ατιμωτική και εξευθυλιστική και κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και συμφωνώ με τα σχόλια της κυρίας Βαλενθιάνο, της Πρόεδρου της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στην Ευρώπη συχνά πιστεύουμε ότι είναι κάτι επιχειωμένο και μεσαιωνικό η θανατική ποινή και θεωρούμε ότι έχει καταργηθεί. Και όμως ε, συνεχίζουμε να έχουμε στενές εμπορικές σχέσεις με χώρες που εφαρμόζουν τη θανατική ποινή σχεδόν καθημερινά. Επίσης ήθελα να σας υπενθυμίσω μια χώρα, δεν θα έλεγα γειτονική ή φιλική, η χώρα εταίρο, τις Ηνωμένε Πολιτείες ε, της Αμερικής, από την οποία έχουμε αντιγράψει την οικονομική πολιτική. Μια χώρα που μας επηρεάζει σε κάθε άποψη και πολιτική. Οι Ηνωμένε Πολιτείε εξακολουθούν να εφαρμόζονται θανατική ποινή. Απίστευτο και όμω αληθινό. Δεν μπορούμε, μάλιστα, ούτε καν να απαιτήσουμε από μια φίλη χώρα όπω είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε να καταργήσει τη θανατική ποινή. Ευχαριστώ κύριε Κοράο και συγχαρητήρια για την αποστολή σας στην Κυριαζία εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δέχεστε μια μπλε κάρτα από τον κύριο Κόρβιν Μίκια, μήπω. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι θα είχε πιο ενδιαφέρον να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Στάνισλαφ Πόλτσακ. Για μισή λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω που μου δίνετε το λόγο στα τσεχικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πρώτο στατή στην προσπάθεια αυτή κατάργηση ανατικής ποινής. Και θα πρέπει πραγματικά να αποτίσουμε ένα φόρο τιμής στις προσπάθειες που καταβάλλονται. Δεν ακούσαμε εδώ επιχειρήματα υπέρ της θανατικής ποινής, γιατί είναι η χειρότερη πράξη βαρβαρότητας που μπορεί κανείς να διανοηθεί. Ακόμα και κατά των εγκληματιών. Επίσης, δεν έχουν μειωθεί τα εγκλήματα από τότε που υπάρχει η θανατική ποινή. Δεν είναι αποτρεπτικός παράγον. Καλό θα ήταν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταφέρει να επιβάλλει παντού δικαιοστάση, αλλά αυτό είναι μια υπόθεση μακράς πνοής. Υπάρχουν ακόμα χώρες που εκτελούν τις θανατικές ποινές. Είναι ε, πολύ σημαντικό τουλάχιστον να επιμείνουμε να υπάρχουν κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές. Δηλαδή, να μην ε, έχει αναδρομική ισχύ η καταδίκη και οι άνθρωποι που εκτελούνται να μην είναι ποτέ ανήλικοι, ας πούμε, εφόσον εκτελούνται. Ή οι γυναίκες έγκυες, ή οι άνθρωποι με αναπηρίες. Και βεβαίως να υπάρχουν ε, αδειάσει τα στοιχεία αποδεικτικά. Ο Πρωθυπουργό Φίτσο έχει εκδώσει ένα βιβλίο ακριβώς ε, με τίτλο «Θανατική ε, ποινή» και σας το συνιστώ, διότι ε, περιγράφει μία σειρά καταστάσεων στις οποίες πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Ευχαριστώ. Η κυρία Αναγκόμες. Ε, και εγώ εστερνίζομαι πλήρω στην άποψη τη Έλενα Βαλεσιάνα, τη ε, Πρόεδρου τη Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Με το ψήφισμα αυτό διατρανώνουμε τη δέσμευσή μα για την κατάρριξη τη θανατική ποινή παγκοσμίω. Ε, ενώ Ιράν, Κίνα και Σαουδική Αραβία είναι χώρε που πρωτοστατούν στι θανατικέ καταδίκε. Εφαρμόζονται μάλιστα θανατικές εκτελέσεις και για τρομοκρατία και για εγκλήματα που συνδέονται με τα ναρκωτικά σε χώρε χωρίς δικονομικέ εγγύησει και πολλές φορές σε δίκες με πολιτικά κίνητρα, όπως συμβαίνει στην Κίνα, κατά Ιγουάρων ή στο Πακιστάν ή στην σημερινή Γουινέα. Και λυπούμε λοιπόν, είναι ντροπή που ανήκει στην κοινότητα των Πορτογαλόφωνων χωρών. Έχουμε λοιπόν πολλές χώρες που εφαρμόζουν θανατική ποινή και προσπαθούμε με την οικονομική υποστήριξη για την καταπολέμηση των ναρκωτικών ε, ουσιαστικά δεν βοηθούμε να καταπολεμηθεί η θανατική ποινή. Και θα πρέπει η στήριξη για την καταπολέμηση των ανθρωπίνων ναρκωτικών να δίνεται στις τρίτες χώρες μόνο εφόσον καταργήσουν τη θανατική ποινή γιατί τελικά οι πολιτικές μας έχουν στήματα τους πιο ανήμπορους στην αλυσίδα ε, των, ε, του λαθρεπορείου ναρκωτικών. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τις πιέσεις ε, στη φαρμακοβιομηχανία που όλο και επινοεί νέα ναρκωτικά που χρησιμοποιούνται σε τρίτες χώρες όπως στις ΗΠΑ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Στάκης Χατζηγεωργίου. Κύριε Πρόεδρε, μόλις προχτές ανακοινώθηκε στη Σαουδική Αραβία ότι θα αποκεφάλιζαν ένα νέο και μετά θα τον σταύρωναν σε δημόσια θέα. Αυτό δεν αποτελεί μόνο προσβολή για τη Σαουδική Αραβία, αποτελεί προσβολή για όλους εμάς που μπορεί να αντιτιθέμεθα, αλλά οι κυβερνήσεις μας και η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά δεν κάνει τίποτα πέρα από ρητορίες. Στο Ιράν κρεμάζουν στους ανθρώπους δημόσια τους κρεμάζουν πάνω στις, ε, στους γερανούς σε δημόσια θέα. Αλλά την ίδια ώρα η κυρία Μογκερίνη επισκέφθηκε τον ηγέτη του Ιράν και δεν μπόρεσε να ψελίσει δύο λέξεις για τις καταδίκες. Στάθηκε μόνο στα οικονομικά συμφέροντα που προκύπτουν και της άρσης των κυρώσεων εις βάρος του Ιράν. Άρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να απαιτήσουμε από τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πούν από αυτό το πράγμα στους ηγέτες αυτών των φορών, να το φωνάξουν και όταν ο κύριος σουλτ θα επισκεφθεί αύριο το ιράν να μην σταθεί μόνο και αυτός στα θέματα των συμφερόντων των οικονομικών να σταθεί και σε αυτά αλλά να ψελίσει δύο κουβέντες για την παραβίαση την αισχρή αυτή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. και μια τελευταία φράση οι ηνωμένες πολιτείες που εφαρμόζουν αυτή τη μέθοδο μειώθηκε καθόλου το έγκλημα στις ηνωμένες πολιτείες; Ευχαριστώ. Ε, Κυρία Ντότς, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Όπως είπαν και πολλοί ομιλητές, το Σάββατο θα υψωθούν πολλές φωνές σε όλο τον κόσμο κατά της θανατικής ποινής και για πρώτη φορά η στήριξη θανατικής ποινής, ε, για πρώτη φορά φέτος στην Ηνωμένο έχει πέσει κάτω από το 50%. Το σημειώνω με χαρά. Θα πρέπει όλοι να συνεχίσουμε να καταδικάζουμε τις χώρες που χρησιμοποιούν πιο πολύ τη θανατική ποινή. Και θα ήθελα, όπως και οι συνάδελφοι, να μιλήσω εδώ ιδιαίτερα για το Ιράν. Και χαίρομαι που οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, Ιράν... Ε, εξομαλύνονται. Αλλά θα πρέπει να έχουμε και δημόσια καταδίκη της κλιμάκωσης χρήση θανατικής ποινής υπό τον πρόεδρο κ. Ροχάνη στο Ιράν. Και είμαι απογοητευμένη που κανείς από τους συντηρητικούς του Ηνωμένου Βασίλειου δεν είναι στην αίθουσα σήμερα για τη συζήτηση. Στο παρελθόν πολλές φορές άφησαν να γίνει η ψηφοφορία κατά συνείδηση στην ομάδα τους. Αποχή πολλές φορές έχουν προτείνει σε τέτοιου είδους ψηφίσματα και ελπίζω πως λόγω της μαζικής χρήση θανατικής ποινής κάποιων μη δημοκρατικών καθεστώτων στον κόσμο θα αλλάξουν αυτή τη στάση του την εβδομάδα στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Εντουάρ Μαχτά. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σχεδόν ομόφωνα εδώ οι παρόντες βουλευτές καταδικάζουμε τη θανατική ποινή. Είναι απάνθρωποι, ε, βα, ε, βάρβαροι, ε, απαξιωτικοί, δεν αρκούν ε, τα κοσμητικά. Δεν πρόκειται ποτέ να είναι αρκετά αυτά. Το είπαν και πολλοί συνάδελφοι. Ε, Παρ' όλα αυτά, ε, ο κατάλογο είναι ακόμα μακρύ των χωρών που σκοτώνουν. Εδώ στην Ευρώπη θα πρέπει να επαγρυπνούμε απέναντι σε λαϊκιστέ που θα του άρεσε ε, να υπάρχει θανατική ποινή ω πανάκια για όλα τα δεινά τη κοινωνία. Όλοι έχουμε στο μυαλό μα τον Ταλή Αλμύρ, 21 ετών που τον συνέλαβαν γιατί συμμετείχε σε μια ε, πορεία για τη δημοκρατία. Δεν πρόκειται εδώ να σας περιγράψω ε, τον ιδεχθή βασανισμό, ε, αλλά να σας πω πόσο θαυμάσια αυτή είναι η προσπάθεια αυτή της νεολαίας που αγωνίζεται για μια πιο δίκαιη και δημοκρατική κοινωνία και μια που είναι παρόν εκπρόσωπο Συμβουλίου. Τελειώνω και τον ερωτώ. Είναι έτοιμο το Συμβούλιο να αγωνιστεί για τον Αλή, για τη δημοκρατία, για τη ζωή κατά της βαρβαρότητας. Θα επιβάλλει στον εαυτό του ως κανόνα της διεθνούς διαπραγμάτευσης, το σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή, το δικαίωμα στη ζωή, αντί για το εμπόριο των όπλων. Ευχαριστώ. Okay. Um... Ευχαριστώ. Και τώρα. Ε, Τσάμπα Μόλναρ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα και κατακτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι έχουμε καταργήσει τη θανατική ποινή όχι μόνο στα κράτη-μέλη της Ένωσης, αλλά και σε πολλά άλλα ευρωπαϊκά κράτη που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι έχει σημασία η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να είναι πρωτοπόρος στην ε, καταπολέμηση θανατικής ποινής. Υπάρχουν χώρες εκτός της Ευρώπης που εξακολουθούν να την επιβάλλουν και να εκτελούν θανατικές ποινές. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τις αποτρέψουμε. Στο παρελθόν, αυτό ήταν ε, και ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτημα, διότι ε, πρόσφατα ο Βίκτορ Όρμπαν, ο Πρωθυπουργό τη Ουγγαρία, άρχισε λέει, να σκέφτεται να βάλει ξανά τη θανατική ποινή. Αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι κατά του ευρωπαϊκού πολιτισμού και η ευρωπαϊκή κοινότητα εξεγέρθηκε για να διατρανώσει ότι είναι πολύ σημαντικές οι αρχές και αξίες μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει παντού ε, να το τονίζουμε αυτό και προς ένα κράτος μέλος, αν μπαίνει σε αυτό τον ολιστήρο δρόμο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στη διαδικασία Catch the τώρα. Ο κύριος Στέτινα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, κατά την Πρωθυπουργία του Ρουχάνη που βουτήθηκε είναι μετριοπαθής, περίπου 2.000 άνθρωποι απαχωνίστηκαν. Με βάση τα στοιχεία της Διεθνούς Αμνηστίας, κατά το πρώτο εξάμεινο του χρόνου, 700 άνθρωποι εκτελέστηκαν και μάλιστα ε, θα περάσουμε τους χίλιους ε, πριν τα τέλη του έτους. Έχουμε τον μεγαλύτερο αριθμό κατακεφαλήν εκτελέσεων παγκοσμίως. Και όσο μιλούμε, ο κύριος Σούλτς ε, πετάει στην Τεχεράνη που θα έχει συναντήσει το Σαββατοκύριακο. Κατά το, τη σύναψη της ε, πυρηνικής ε, συμφωνίας με το Ιράν δεν θα πρέπει να ξεχνούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Φροντζούλικα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, με ισχύει ιδιαίτερα το γεγονός ότι σε αντίθεση με τις γενικές τάσεις των τελευταίων δεκαετιών, όλο και περισσότερες χώρες θέσπισαν νομοθεσίες που επιτρέπουν τη θανατική ποινή για εγκλήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά. Ε, στηρίζω την έκκληση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, να συμπεριλάβει την εκστρατεία της εξωτερικές σχέσεις και στην εξωτερική πολιτική για να καταργηθεί η θανατική ποινή και επίσης να εντατικοποιηθούν ε, οι συνοπηλίες με χώρες που αυξάνουν τον αριθμό των εκτελέσεων ή επαναφέρουν την θανατική ποινή. Είναι απάνθρωπη, ατιμωτική, επαξιωτική και εξευτελιστική τιμωρία η θανατική καταδίκη και απειλεί τη θανατικη ποινη ειναι απανθρωπη ατιμωτικη απαξιωτικη και ξεφτυλιστικη τιμωρια ζωή που κατοχυρώνεται στην Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πρόκειται για μία πράξη βασανιστηρίου απαράδεκτη για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει να διατρανώσουμε τη θέση μας κατά της θανατική ποινή και να προβλέψουμε οικουμενικό δικαιοστάσιο της θανατικής ποινή προκειμένου ε, κάποια στιγμή να καταργηθεί πλήρω και αυτό να αποτελέσει βασικό στόχο της πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστούμε κύριε Ευρωβουλευτά. Ο κύριος Νότης Μαριάς τώρα. Κύριε Πρόεδρε, όλα τα κράτη της Ένωσης έχουν πλέον καταργήσει τη θανατική ποινή, καθώς η κατάργησή της αποτελούσε προϋπόθεση για την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση η θανατική ποινή όμως συνεχίζει να εφαρμόζεται σε χώρες όπως οι Ηνωμένε Πολιτείε, η κίνα και σε πολλά κράτη του μουσουλμανικού κόσμου όπως η σαουδική αραβία και το ιράν. το δικαίωμα στη ζωή δεν θα πρέπει να αφαιρείται από κανένα και με κανένα τρόπο. οι ποινές που επιβάλλονται σε κάποιο κατηγορούμενο κατόπιν δίκαιης δίκης πρέπει να έχουν αφενός σοφρονιστικό και αφετέρου αποτρεπτικό χαρακτήρα με βάση αυτέ τι αρχέ, είναι απαράδεκτη η στάση συγκεκριμένων κυβερνήσεων οι οποίε προτείνουν ανοιχτά ή συγκαλυμμένα την επαναφορά τη θανατική ποινή, αμφισβητώντα έτσι τον σεβασμό τη ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα. πρέπει όμω για συγκεκριμένα ή δεχθή εγκλήματα ή αδικήματα να επιβάλλονται βαρύτατες ποινές οι οποίες να έχουν παραδειγματικό και αποτρεπτικό χαρακτήρα χωρίς όμως να φτάνει κανείς στην επιβολή της εσχάτης των ποινών που είναι η δεχθεί εγκληματα η αδικηματα να επιβαλλονται βαρυτατε ποινε οι οποιε να εχουν παραδειγματικο και αποτρεπτικο χαρακτηρα χωρι ομω να φτανει κανει στην επιβολη τη εσχατη των ποινων που ειναι η επιβολη τη θανατικη ποινη τάσσομαι λοιπόν υπέρ της πάυσης της θανατικής ποινής σε ολόκληρο τον κόσμο. Η θανατική ποινή προσβάλλει την αξία του ανθρώπου μετατρέποντας τον κατάδικο σε αντικείμενο με σκοπό τον παραδειγματισμό και ακυρώνει την ίδια την έννοια των δικαιωμάτων του ανθρώπου αφού τερματίζει πρόωρα την ανθρώπινη ιδιότητα. γι' αυτό άλλωστε η θανατική ποινή έχει απαγορευτεί σύμφωνα με το δεύτερο πρωτόκολλο του διεθνούς συμφώνου του οργανισμού ηνωμένων εθνών για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα όπως και με σειρά άλλων κειμένων του διεθνούς δικαίου. η ευρωπαϊκή ένωση θεμελιώνεται πάνω στις αξίες της προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων και αποσκοπεί στην προώθηση αυτών ακριβώς των αξιών σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 της ιδρυτικής της συνθήκης. Συνεπώς, η Ένωση οφείλει να προωθήσει με μεγαλύτερη ενεργητικότητα την κατάργηση της θανατικής ποινής στις χώρες με τις οποίες συναλλάσσεται σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο. Πρέπει να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να τερματιστεί οριστικά αυτή η βαρβαρότητα. ευχαριστώ. Ε, ο κύριο Σόλτες έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Περί τίνος πρόκειται εδώ. Είναι ένα θέμα ε, στο οποίο θα πρέπει πάντα να επαγρυπνούμε. Η ε, επιβολή της θανατικής ποινής είναι ε, μια πράξη κατά του πολιτισμού και εμείς πρέπει πάντα να την αποκρούμε και να αγωνιζόμαστε για την κατάργηση. Ε, το δικαίωμα στη ζωή είναι αναπαλωτρίωτο. Τα κράτη που επιβάλλουν θανατική ποινή μπορεί να ε, καταδικαστούν και πρέπει να καταδικαστούν ε, δημόσια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δυνατότητες να το κάνει αυτό και να ασκήσει πολιτική πίεση με τα οργανά της και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι σωστό αυτό ε, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύεται συμφωνίες με διάφορες χώρες θα πρέπει να θέτουμε υπόψη ε, αυτό το ζήτημα και να καλούμε τις χώρες να καταργήσουν τη θανατική ποινή με επιχειρήματα και να μην υπογράφουμε τελικά συμφωνίες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μπάτον έχει το λόγο. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η προφορική ερώτηση ζητεί από το Συμβούλιο να ασκήσει πίεση στις χώρες αυτές που ακόμα επιβάλλουν τη θανατική ποινή για να την καταργήσουν. Θα απαντήσει το Συμβούλιο ότι δεν κάνει τίποτα γιατί αδιαφορεί απολύτως. Η ε, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να πει σε πολιτισμένα κράτη ε, ότι δεν μπορούν να εκτελούν τους χειρότερους εγκληματίες. Και μιλώ για εγκληματίες, όχι για πολιτικούς αντιφρονούντες. Υπάρχουν ε, ε, δολοφόνοι διάφοροι διαβόητοι που θα πρέπει να πληρώσουν για τα εγκλήματά τους με τη ζωή τους. Γιατί όχι. Αν αύριο γίνει δημοψήφισμα στην Αγγλία για την επιστροφή της εισχάτης των ποινών. Υποθέτω ότι θα την υπερψηφίσουν οι Βρετανοί και εγώ οπωσδήποτε. Ελπίζω αυτά τα πολιτισμένα κράτη που έχουν ε, την θανατική ποινή θα πούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην ανακατεύεται στα θέματα τους και να κοιτάει τη δουλειά της. Ευχαριστώ. Κύριος Ξύπ. Πριν σας δώσω το λόγο κύριε Ξύπ, θα ήθελα να διευκρινίσω σε, όσο, σε όλους όσους ζήτησαν το λόγο σε αυτή τη διαδικασία ότι με βάση ε, τον κανονισμό πρέπει να έχουν δηλώσει ε, ότι θέλουν να λάβουν το λόγο στο ΚΑΤΣΔΙ πριν ξεκινήσει η σχετική συζήτηση. Αλλιώ δεν δικαιούνται να λάβουν το λόγο. Κύριε Ξύπ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κάθε χρόνο έχουμε την συζήτηση αυτή για συγκεκριμένο λόγο, γιατί πιστεύουμε ότι κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στη ζωή. Αυτό το δικαίωμα είναι αναπαλωτρίωτο και θεμελιώδες ε, ανθρώπινο δικαίωμα. Προκύπτει από το φυσικό δίκαιο και από την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός πέρασε μια εποχή που εφαρμοζόταν ε, ε, η θανατική ποινή, ακόμη και σε ευρωπαϊκές χώρες. Εγώ κατάγομαι από μια χώρα που πριν από 25 χρόνια εφάρμοσε δικαιοστάσιο και τελικά κατήργησε τη θανατική ποινή. Το θέμα είναι, έχουμε μέσα στη διάθεσή μας για να καταργήσουμε τη θανατική πίνη σε όλες τις χώρες. Αυτή είναι μια διαδικασία καθόλου εύκολη. Γιατί πάντα υπάρχουν σοβαρά επιχειρήματα που προτάξουν, προτάσουν οι συνομιλητές μας που δεν θέλουν να καταργήσουν τη θανατική πίνη. Για παράδειγμα, ότι έχει αποτρεπτικό χαρακτήρα, ότι υπάρχουν σοβαρά εγκλήματα όπως η τρομοκρατία που πρέπει να τιμωρούνται έτσι. Και μάλιστα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε υιοθετήσει πολλά ψηφίσματα που ζητούν ε, άνθρωποι που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο να απελευθερωθούν, ιδιαίτερα όταν έχουν καταδικαστεί για πολιτικούς λόγους. Ε, και το έχουμε πετύχει. Και αυτό είναι σημαντικό στοιχείο της πολιτικής που ασκούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που επιδιώκουμε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Κατερίνα Τσινίτσι έχει το λόγο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κατάργηση της ε, θανατικής ποινής ήταν ένα από τα σημαντικά επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε όμως εκατοντάδες ε, εκτελέσεις το τελευταίο χρόνο σε πάνω από 20 χώρες. Θα πρέπει λοιπόν ε, με αποφασιστικό τρόπο να συνεχίσουμε την αποστολή μας για να καταργηθεί η θανατική ποινή παγκοσμίω. Η ανθρώπινη ζωή και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι οικουμενικές αξίες και θα πρέπει να τις υπερασπίσουμε με κάθε ειρηνικό μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας. Θα πρέπει να ασκήσουμε ε, στεναρή πίεση στις χώρες και στις κυβερνήσεις που εφαρμόζουν τη θανατική πίνη και να προβλέψουμε πιο αποτελεσματικά γενικότερα μέτρα για νομοθετική μεταρρύθμιση και φυσικά να μπλοκάρουμε την εκτέλεση θανατικών ποινών με νομοθετικά μέτρα ή να αποφύγουμε την, ε, ε, τις θανατικές καταδίκες δεν θα πρέπει το αίτημα για κατάργηση θανατική ποινής να θεωρείται ως πολιτιστική επικιοκρατία ή επέμβαση στα εσωτερικά μιας χώρας. Η θανατική μια χωρας είναι άδικη. Γι' αυτό και η ανοχή μας απέναντί της θα πρέπει να είναι μηδενική. Ευχαριστώ. Ο κύριο Κάσκη έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Η ανθρώπινη ζωή είναι η σημαντικότερη αξία Γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι έχουμε διαφορετικές καταστάσεις ε, που οδηγούν στην ε, ε, θανατική ποινή. Και σε όλες τις περιπτώσεις είμαστε κατά της θανατικής ποινής. Αυτό το ακούσαμε στη διάρκεια της συζήτησης. Ακόμη και για δολοφονίες, ακόμη και για τα ιδεχτέστερα έγκληματα, ε, το διεθνέ δίκαιο είναι κατά τη θανατικής ποινή. γι' αυτό και φροντίζουμε, προσπαθούμε οι χώρες σταδιακά να το καταργήσουν, ακόμα και αυτές που το έχουν ακόμη, γιατί πρόκειται για μια απερχαιωμένη τιμωρία. Όμω έχουμε και μια άλλη του κατάσταση. Έχουμε την α, θανατική ποινή για εγκλήματα που συνδέονται με τα ναρκωτικά, για μοιχεία και ούτω καθεξής. Ε, μάλιστα, η οι θανατικές αυτές ποινές είναι ουσιαστικά δικαστικά εγκλήματα. Είναι αναφυσβήτητο ότι οι συγκεκριμένοι δικαστές ε, που επιδικάζουν αυτές τις ποινές ε, είναι οι ίδιοι δικαστές εγκληματίες. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Γερμανοί ναζιστές ε, δικαστές επίσης προσήχθησα στο δικαστήριο και πιστεύω ότι θα πρέπει να σύρουμε στα δικαστήρια τους δικαστές που ε, εκφωνούν καταδικαστικές αποφάσεις για θρησκευτικά εγκλήματα, για εγκλήματα που συνδέονται με ναρκωτικά ή για εγκλήματα που με βάση την οικουμενική δικαιοδοσία δεν δικαιοδοσία σε καμία περίπτωση να τιμωρούνται με τέτοια ποινή. Ευχαριστώ κυρία Λίνα Μπέλαν. Πολύ χαιρετίζω τη συζήτηση που γίνεται για τη θανατική ποινή, γιατί είναι μια ευκαιρία για μας να αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει μεγάλη αντίδραση από τα ευρωπαϊκά κράτη για το θέμα αυτό. Αλλά θα ήθελα να σκεφτούμε τον Ιμπραχήμ Χαλάουα, έναν Ιρλανδό έφηβο που είναι ο μοναδικός Ευρωπαίος που είναι σε Αιγυπτιακή φυλακή από το καλοκαίρι του 2013 και που απειλείται με τη θανατική ποινή. Και γιατί, γιατί πήγε σε μία διαδήλωση και η Διεθνής Αμνηστία λέει πως η φυλάκισή του είναι κατά του άρθρου, παραβιάζει το άρθρο 2 της συνθήκης Euromed. Χαίρομαι λοιπόν για τα όσα είπε ο κύριος Σμιτ σήμερα. Θα πρέπει να είναι πιο βροντερή η φωνή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το θέμα αυτό. Πράξεις, όχι λόγια, η Αίγυπτος είναι έβδομη στον κατάλογο των θανατικών ποινών και νομίζω πως έφτασε η ώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την Ιρλανδική κυβέρνηση να δράσουν εναντίον της Αιγύπτου έτσι ώστε οι διάφοροι Ιμπραχήμ Χαλάι που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη φυλακή και περιμένουν να εκτελεστούν να σωθούν. Ο κύριος Καστάλντο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Στις 2 Οκτωβρίου εορτάσαμε την Διεθνή ημέρα κατά της θανατικής λυπηρή ημέρα γιατί η θανατική Είναι μία ακόμα λυπηρή ημέρα γιατί η θανατική ποινή ζει και θριαμβεύει. Ξέρετε πως υπάρχει μια μεγάλη ομάδα κρατών που στηρίζει αυτό το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Η Ιαπωνία, η ΙΠΑ και στρατηγική σύμμαχοι, η Αίγυπτος, το Πακιστάν, η Σαδική Αραβία, η Λευκορωσία, που είναι δύο βήματα από την Ευρώπη, που χρησιμοποιούν αυτό το την αποτρόπια πρακτική για να προχωρήσουν σε κάθαρση των πολιτικών αντιπάλων που έχουν το θράσος, να φέρουν αντιρρήσεις και να αντιδρούν. Σχέσεις μας με το Ιράν. Δεν μπορούμε να δώσουμε την επόμενη λευκή επιταγή γιατί η εμπορική σχέση είναι βασικό εργαλείο για να προχωράμε και στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 700 καταδίκες σε θανατική ποινή στο Ιράν, 2.200 στην Κίνα, που είναι ένας μεγάλος εταίρος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πότε θα χρησιμοποιήσουμε πια την οικονομία και το εμπόριο ω ένα εργαλείο για να γίνουν σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και να μην γίνεται το αντίστροφο. Γιατί εμεί είμαστε η Ευρώπη, να παραμείνουμε η Ευρώπη, να συνεχίσουμε τη μάχη κατά αυτή τη ποινή και να καταδικάζουμε τι σημαίνει η θανατική ποινή. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Ρούζα Τόμασιτ. Ευχαριστώ. Η Ευρώπη έχει τη θέση της ε, για τη θανατική ποινή και είναι σχεδόν ομόφωνη. Ε, είμαι ιδιαίτερο ευτυχή ε, που οι κοινωνίε μα ε, ξεπέρασαν και κατήργησαν αυτή την απειρχιωμένη μέθοδο και ακόμη και στα, απέναντι στα δεχτέστερα εγκλήματα συμπεριφερόμαστε όπω ταιριάζει σε ανθρώπου που ο πολιτισμό του διαμορφώθηκε από τη χριστιανοσύνη. Θεωρώ ότι την άποψή μα θα πρέπει να το προωθήσουμε και στον υπόλοιπο κόσμο, κυρίω στι σχέσει μα με τρίτε χώρε με τι οποίε έχουμε στενού εμπορικού, οικονομικού, διπλωματικού ή στρατιωτικούς δεσμούς. Θα πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη και τις πολιτιστικές, ε, πολιτισμικές συγγνώμη, διαφορές και αυτή την ε, ε, δύσκολη και λεπτή πολιτική στιγμή να διαλέξουμε με τι μέσα θα προωθήσουμε την κατάρριση της θανατικής ποινής που πραγματικά δεν έχει θέση στον 21ο αιώνα. Ευχαριστώ. On behalf of... Uh, εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το λόγο έχει ο Επίτροπος κύριος Σμιτ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, για να ολοκληρώσουμε θα συμπεράνω ότι η θανατική ποινή δεν έχει θέση τον 21ο αιώνα. Σας ευχαριστώ για την ευρύτατη ε, και στεναρότατη προσήλωσή σας ενάντια στη θανατική ποινή. Και αυτό είναι και ένα σαφέστατο μήνυμα που θα πρέπει να εκπέμψουμε προς τις χώρες οι οποίες ακόμα δεν έχουν προσγειωθεί στον 21ο αιώνα όπως το είπατε. Δεν υπάρχει εύκολη λύση. Είναι προφανές ότι σε κάθε ευκαιρία θα πρέπει να χρησιμοποιούμε την πυθό, να συζητούμε, να κινητοποιούμε ε, την κοινωνία των πολιτών μας, τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις μας, έτσι ώστε πραγματικά να επιτεθούμε σε αυτή την πρακτική άλλων εποχών. Η διεθνής ε, κοινή γνώμη μπορεί επίσης να διαδραματίσει πολύ σπουδαίο ρόλο. Και εδώ σκέφτομαι όλα αυτά που γίνονται στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών. Βεβαίω είναι πάρα πολύ μακροσκελή αυτή η διαδικασία γιατί στο μεταξύ χιλιάδε άνθρωποι εκτελούνται. Αλλά πιστεύω ότι ε, φαίνεται από τη συζήτηση που κάνουμε σήμερα ότι η Ευρώπη εδώ είναι πιστή στι αξίε τη. Οι αξίε αυτέ θα πρέπει να γίνουν ακουστέ και στις χώρες που δεν ε, τις ημερίζονται. Μα το γράφουμε, έχουμε και τις διάφορες συμφωνίες που περιλαμβάνουν ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στι συμφωνίες με τις χώρες. Θα πρέπει όμως να είμαστε και ρεαλιστές. Δεν μπορούμε ε, σήμερα να οδηγήσουμε σε εμπλοκή ή να τιμωρούμε ε, απορρίπτοντας κάθε συμφωνία με χώρες που εκτελούν θανατική ποινή. Γιατί αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Δια του διαλόγου καλύτερα και με πολύ σαφή μηνύματα θα ε, ε, τους κάνουμε να αλλάξουν και παραμένουν αισιόδοξου ότι κάποια στιγμή θα προσγειωθούν οι χώρες αυτές στον 21ο αιώνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Υπουργέ. Ολοκληρώνουμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό.